per Επίσης ε, υπάρχει αίτημα για την άρση της ασυλίας ε, της κυρίας Ρολάντα Πάξας ε, στο πλαίσιο μιας δικαστικής αγωγής. Αυτό το αίτημα παραπέμφθηκε στην Επιτροπή, Νομική Επιτροπή του Κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για